Right, good morning, ladies and gentlemen. It's minutes. Καλημέρα σας. Είναι 9 και 3 λεπτά. Να αρχίσουμε την κοινή μας συνεδρίαση. Σας παρακαλώ καθίστε. Και όσοι πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσουν να συζητούν μεταξύ τους, παρακαλώ να βγουν έξω. οι πράσινοι κάνουν θόρυβο. Λοιπόν, από πλευράς της ε, κυρίας ε, Προέδρου της Επιτροπής Πολιτισμού και μου, καλώς ήρθατε στην κοινή συνεδρία των δύο επιτροπών μας, της ΑΦΕΤ και της ΚΟΥΛΤ. Και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία για το σχέδιο έκθεση προς μια στρατηγική της Ένωσης για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις. Πρώτα απ' όλα να ρωτήσω τους εισηγητές αν θέλει κάποιος να πει κάτι. Μου είπαν ότι δεν έχει έρθει ακόμη ο κύριος Μπροκ. Μήπως η κυρία Σιλβία Κώστα θέλει να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε. Θα συνεχίσω Ιταλικά, παρακαλώ. Να ευχαριστήσω Θέλω να εκφράσω τη χαρά μου και την ικανοποίησή μου για αυτή τη σημαντικότατη έκθεση που ετοιμάσαμε για την ανακοίνωση. Τη θεωρούμε στρατηγική σημασία και θέτει μια θεώρηση πιο ολοκληρωμένη, πιο σφαιρική για τις πολιτιστικές σχέσεις σε διεθνές επίπεδο. Να θυμίσω ότι το Κοινοβούλιο το 2011 ήταν το πρώτο όργανο που οδήγησε προς αυτή την κατεύθυνση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μια σχετική έκθεση μια προπαρασκευαστική δουλειά που είχαμε ετοιμάσει στις Επιτροπές Πολιτισμού, στην Επιτροπή Πολιτισμού τότε. Χαίρομαι πολύ λοιπόν που αυτή η σχέση συνεργασία έχει οδηγήσει σήμερα σε αυτό το αποτέλεσμα με τη συνεργασία και του τότε Πρόεδρου Μπροκ και να ευχαριστήσω και όλους τους σκιώδεις εισηγητές ε, για μία ενιαία στρατηγική που βεβαίω δεν ξεκινάει σήμερα τα πρώτα βήματα, αλλά ήδη έχει κάνει πολλέ ε, έχει επιτελέσει πολλά βήματα προόδου στο επίπεδο των πολιτιστικών σχέσεων, αλλά στο επίπεδο του διαπολιτιστικού διαλόγου, την προώθηση του πολιτιστικού, της πολιτιστικής κληρονομιάς ε, και σε σχέση με τρίτες χώρες. Τα σχετικά οικονομικά ωφέλη, λόγω χάρη τον ε, τομέα των οπτικοακουστικών και της δημιουργίας, των δημιουργών, όλα αυτά ε, πρέπει να προωθηθούν. Χρειάζεται και ο πολιτισμό ω τέταρτο πυλώνα τη βιώσιμη ανάπτυξη και εμεί, ε, οι δύο επιτροπέ μαζί, δείξαμε πόση σημασία δίνουμε σε αυτή τη διάσταση. Σα ευχαριστώ πολύ για την τόσο θετική συνεργασία. Ευχαριστώ και τι γραμματείε των δύο επιτροπών, του πιο συζητητέ, όλου μα του ε, συνεργάτε και όσου συνεργάστηκαν στο θετικό αυτό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν άλλα σχόλια. Όχι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Τροπολογία 80. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στην 91. Παρακαλώ. Πώς είπε. Ο κύριος Νέκοφ λέει ότι δεν μπορεί να ψηφίσει. Δεν λειτουργεί το μηχάνημα ψηφοφορίας του. Α, τώρα λειτουργεί. Α, ωραία λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν, τροπολογία 91 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Περνάμε στην παράγραφο 5. Υπέρ. Συγγνώμη, είναι συμβαστική. 6. Ωραία, με συγχωρείτε. Εντάξει, θα ξυπνήσω. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Καλώς. Ψηφίζουμε επί της συμβαστικής 7. Κύριε Πρέτα, δεν έχουμε χρόνο για αστεία. Ωραία. Πέρας. Α, καλά που το ελέγξαμε. Συμβαστική 7 ενεκρίθη. Οπότε περνάμε στη συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα να πάμε στην 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 128 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 130 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 129 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 139 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 134 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 136 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 138 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται, συγγνώμη. 137 κατά τμήματα. Το πρώτο τμήμα παρακαλώ, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 139 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 140-141 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 143 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 142 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 144 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 145 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 146 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε στην 148 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 149 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 155 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 156 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 163 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 169 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 170 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 172 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 173 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 176 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 174 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 175 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 183 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε έτσι ώστε να ξυπνήσουμε κιόλας 183 άρχεται πέρας απορρίπτεται. Υπέρ 33 κατά 39. Αυτή ήταν 183. Απορρίπτεται. Έχουμε τις 184, 5, 6 και 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 188 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 190 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 192 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 191 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 200 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 203 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 204 υπέρ κατά αποχές Ας ελέγξουμε. Τη 204. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 206 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 207 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 205 υπέρ κατά εποχές ας ελέγξουμε. Ε, συγγνώμη, 208. 208 ψηφίζουμε. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην συμβαστική 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2.18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 220 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.37 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε. 2.37 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 2.38 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 2.39 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 2.44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 2.45 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 2.46 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 2.48 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 2.47 υπέρ, να ελέγξουμε τη 2.48, καλώς. Ελέγχουμε τη 2.48, άρχεται. Πέρας. Ήταν αρκετά σαφές, όχι. Λοιπόν, 2,47 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 2,49 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 2,51 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 2,50 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 2,52 και 3 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 2.54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 2.65 του κυρίου Χριστέα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2,73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2,74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2,81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2,82 και 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 289 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 286 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Α, συγγνώμη, ούτως ή άλλως καταπίπτει. Ωραία. Οπότε μπορούμε να πάμε στην 285. Θαυμάσιο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 290 και 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 294 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.98, 99 και 300 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 301 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 302 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 303 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 304 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 305 και 6 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτονται. 307 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 308 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 309 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 310 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 311-12 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτονται. 313 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 όχι υπέρ, 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε στην 43 υπέρ κατά αποχές συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Περνάμε 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ κατά αποχές Ας ελέγξουμε την 51 λοιπόν. Άρχεται. Έχουμε 80 συναδέλφους ε, παρόντες, δύο ή μάλλον ένας μόνο, κοιμάται ακόμη. Ένας φαίνεται ότι εξακολουθεί να κοιμάται, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 46 υπέρ 33 κατά. Επί της 51. Τρίπελ. Εγκρίνεται λοιπόν. Λοιπόν, έχουμε την προφορική τροπολογία 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 1 υπέρ. Α, συγγνώμη, κατά πίπτη, συγγνώμη. Οπότε, 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Ωραία, να ελέγξουμε. Την 58. Πέρας. Α, εγκρίθηκε. Ωραία. 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 69 υπέρ κατά αποχές. Ας ελέγξουμε την 69. Άρχεται. Πέρας φορές. Εγκρίθηκε. 41 ψήφι υπέρ, 38 κατά. 70 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 74 υπέρ κατά αποχές. Ας ελέγξουμε την 74 του κυρίου Ράγκελ, Ρανζέλ. Τρεις συνάδελφοι δεν έχουν ψηφίσει ακόμη. Α, δύο. Ένας. Πέρας. 26-53. Απορρίπτεται σαφώς. 73 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 75 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 76 υπέρ, κατά αποχές οι σοσιαλιστές είναι υπέρ ωραία εγκρίθηκε τότε 78 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε το 78 άρχεται η ψηφοφορία πέρας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 απορρίπτεται. 14 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ, 18 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές. Ας ελέγξουμε τη 18. και τη 16. Οι σοσιαλιστές θέλουν να ελέγξουμε πρώτα την 16. Αρχίζουμε λοιπόν με την 16. 16. Πέρας. Εγκρίνεται. Με 40-37. Και τώρα ελέγχουμε την 18. Υπέρ. Κατά αποχές α, α, μισό λεπτό, μισό δεν λειτουργεί το μηχάνημα ένα σφυρί να του δώσουμε μία λοιπόν τι κάνουμε τώρα α τώρα λειτουργεί, ωραία ελέγχουμε τη 18 Δύο συνάδελφοι δεν ψήφισαν ακόμη. Ένας, ωραία πέρας. 46 υπέρ, 33 κατά, εγκρίνεται. Οπότε, πρέπει να υπάρξει και τελική ψηφοφορία. Α, μάλιστα. Οπότε, τελική ψηφοφορία στο σχέδιο έκθεσης συνολικά, ονομαστική, Ένας δεν έχει ψηφίσει ακόμη. Πέρας. Εγκρίνεται 62 υπέρ, 13 κατά και 4 αποχές. Συγχαρητήρια στους εισηγητές. So I now the honor of closing our joint meeting with and in εδώ λίγη η κοινή μας συνέντευξη με την Επιτροπή Κόλτ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, και θα συνεχίσουμε χωρίς τα